Hello everyone. Hello everyone. Καλησπέρα σε όλους. If you wanna take your... Καθίστε παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη για να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίαση. Γιατί ξέρετε κάποιοι από εμάς έχουμε να πάμε και σε τριμερή διάλογο μετά, οπότε θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα να μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τάχιστα. Πολύ ενδιαφέρον υπάρχει. Και χαίρομαι πολύ που είστε πολύ πληθέστατοι εδώ. Ο κύριος Γκουαλτιέρη όμως δεν μπορούσε να είναι εδώ. Εγώ λοιπόν θα προεδρεύσω αυτή τη κοινή συνεδρίαση μεταξύ των Επιτροπών Περιβάλλοντο και Οικονομικών Υποθέσεων, ΛΥΜΠΕ, ΕΚΟΝ. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ψηφοφορία. Πριν από αυτό, θέλω να ξέρω κατά πόσον υπάρχει κάποια αντίρρηση σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη. 19 γλώσσες προβλέπονται σήμερα στο πλαίσιο της διερμηνίας και φυσικά υπάρχει ηλεκτρονική τεκμηρίωση και ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης. Έχουμε τα πρακτικά της 6ης Δεκεμβρίου και της 22ης Ιανουαρίου της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αν δεν έχετε αντίρρηση εκφράσει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, σας θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Αυτά ήταν τα εισαγωγικά και περνάμε στην ψηφοφορία ευθύ αμέσω. Ελπίζω να έχετε έτοιμε τι κάρτε σα, τι κάρτε ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε όμως θέλει το λόγο κυρία Μπερές. Ναι, θέλω να σας πω ότι στο σύνολο δεν έχω μαζί μου την ε, κάρτα μου, οπότε πρέπει να με μετράτε εμένα. Α, δεν ήρθες θα τα προετοιμασμένη, λοιπόν, δεν πειράζει όμως. Θα σημειώνουμε τι ψηφίζεται και θα περάσουμε στην ψηφοφορία για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της θέσπισης πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων. Η κυρία Μπέρις λοιπόν θα ψηφίζει διαχειρός και παρακαλώ η γραμματεία να σημειώνει. Πρόσφατα πρόταση λοιπόν κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων, συμβιβαστική όχι, τροπολογία 124 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική A ψήφι υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Παρακαλώ. And the vote is closed. And it's ναι, ναι. Πέρας. Αποσύρθηκε με μία ψήφο διαφορά. Δεν ξέρω αν βλέπετε το αποτέλεσμα. Το βλέπετε. Κύριε Μπερή, σας ήταν υπέρ ή κατά. Είστε υπέρ. Και πάλι απορρίπτεται όμως σε συμβαστική, γιατί είναι πάλι 53, αλλά 53 όλα. Ψηφ, ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. Πηγαίνουμε τώρα στη συμβιβαστική A2, α2. Ησυχία για να συγκεντρωθούμε. Ψηφίζετε, ξέρετε, πάνω από 100 άνθρωποι εδώ. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Πέραση about ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στη σελίδα 4, ησυχία. Συμβιβαστική B, Β, ψήφι περ. Α, ναι. Υπάρχει προφορική τροπολογία που έχει ζητήσει το ΕΛΚ. Την έχετε στη λίστα. Υπάρχει κάποιος που αντίθετος με την τροπολογία αυτή. Είστε αντίθετοι, ε? Ωραία. Πάνω από 7 είναι αντίθετη που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να την θέσουμε σε ψηφοφορία αυτή την προφορική τροπολογία. Θα ψηφίσουμε τη Β χωρίς την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ λοιπόν συμβαστικής Β χωρίς την προφορική τροπολογία. Κατά, αποχές, νομίζω απορρίπτεται, θα ήθελα όμως να ελέγξουμε. And the vote is... Πέρασε. Ησυχία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία και σχεδόν λίγη. Τώρα έληξε. Εγκρίνεται. Σελίδα 6. Ψηφίζουμε την τροπολογία 315. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 316. Α, είναι ταυτόσιμη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πηγαίνουμε σε βαστική C, ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική CA, ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. CA2. Α, θέλετε να ελέγξουμε τη CA, να την ελέγξουμε, συμφωνώ και εγώ, ας ελέγξουμε. I Έκανα μια απόπειρα να συντομεύουμε, αλλά... Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε πράγματι και περνάμε στη CA2. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική D. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται D2 ψήφι υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται σελίδα 13 τώρα αν τη βρω κι εγώ συμβαστική DA ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική E ε ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F, ψήφι ΠΕΡ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Ναι, ναι, συμφωνώ. Να ελέγξουμε και συμβιβαστική άλλωστε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εσείς είστε υπέρ εγκρίνεται με μία ψήφο. Εντάξει, εντάξει, εντάξει, μη διαμαρτύρεστε. Η κυρία Μπερές είπε την υπέρ. Τι να κάνω εγώ. Ήταν 52 όλα. Συμβαστική F2. Όχι, δεν την ψηφίζουμε. Πού πηγαίνουμε στη σελίδα 17. Συμβιβαστική FA. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές ελέγχου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Από την κυρία Ζόμερ. Ξέχασα να φέρω την κάρτα ψηφοφορίας μου. Είμαι κατά. Στις προηγούμενες ψήφους, ψηφοφορίες, ε, τότε θα πρέπει να ζητήσω να μου πείτε τι ψηφίζετε, υπέρ κατά. Τέλο πάντων, έβλεπα ότι σήκωνε το χέρι, αλλά δεν είχα ζητήσει, δεν τη είχα δώσει το λόγο να μα πει τι ήθελε. Τέλο πάντων. Συμβιβαστική ψηφίζετε Ψηφίστε υπέρ κατά. Order. If, if it's available for... Αν το επιτρέπω σε έναν, θα το πρέπει να το επιτρέψω και σε άλλους. Κύριε Μπέρις, θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο γι' αυτό. Είναι σίγουρα πάρα πολύ λεπτό ε, το να προεδρεύει κανείς, ιδίως σε μια κρίσιμη ψηφοφορία. Όταν λέτε ότι εγκρίνεται ε, μια τροπολογία, ε, η ψηφοφορία ολοκληρώνεται και δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Καταλαβαίνω τι λέτε κυρία Μπερές, λέει πρόεδρος. Αλλά υπάρχει και πολύ θόρυβος. Εσείς έχετε διατελέσει πρόεδρος Σέκον το γνωρίζω και ξέρω πόσο εμπειρίστε. Όμως είδα να σηκώνει το χέρι της η κυρία Ζόμερ πριν. Δεν της έδωσα όμως το λόγο. Γι' αυτό και λέω ότι είναι δίκαιο να της ζητήσω να μας πει τι ψήφισε υπέρ κατά. Αυτό θα ήταν το δίκαιο. Δεν έχουν φέρει όλοι τις κάρτες ε, για να ψηφίσουν και υπάρχει κάποια σύγχυση. Τέλο Τέλος πάντων, είναι δίκαιο να δώσω το λόγο στην κυρία Ζόμερ, γιατί δεν, μάλλον να μας πει τι ψηφίζει η κυρία Ζόμερ, γιατί είχε σηκώσει το χέρι και δεν της έδωσα το λόγο. Να επαναλάβουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Ακούστε, εγώ αποφασίζω, λυπούμε, θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία επί της συμβαστικής F. Και τώρα μπορείτε να ξαναψηφίσετε αλλά θα λάβουμε υπόψη όλες και όλους που δεν έχουν φέρει την κάρτα τους. Ψηφίζουμε ξανά την ΕΦ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Κύριε Μπερές, εσείς τι ψηφίζετε, πρέπει να μας το πείτε, για να λάβουμε υπόψη την ψήφο σας. Εσείς είστε υπέρ. Ποιος άλλος δεν έχει κάρτα ψηφοφορίας, η κυρία Ζόμερ που ψηφίζει κατά, εντάξει, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην FA. No, you have to go to compromise FA. No, if it's Okay. Okay, then we have to... Κυρία Μπερές. Το 178 άρθρο του κανονισμού λέει ότι ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη ψηφοφορίας και τη λήξη ψηφοφορίας. Άπαξ και ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη μιας ψηφοφορίας. Καμία παρέμβαση, ούτε καν ο πρόεδρος δεν επιτρέπει πριν τη λήξη της ψηφοφορίας, αν μπλα μπλα μπλα. Ο πρώτος αποφασίσει. Δηλαδή δεν υπάρχει παρέμβαση, δεν υπάρχει διακοπή μετά την έναρξη ψηφοφορίας. Ε, άρα δεν μπορούσατε, δεν είχατε δικαίωμα να επαναλάβετε την ψηφοφορία ψηφοφορία. Καταλαβαίνω τι λέτε, λέει πρόεδρο, κυρία Μπερές. Αν ε, δεν θέλετε να επαναληφθεί η ψηφοφορία, εγώ απλά ε, έκανα ένα λάθος στην καταμέτρηση, κυρία Μπερές, γιατί δεν μέτρησα την ψήφο της κυρία Σόμερ. Γι' αυτό επανέλαβα την ψηφοφορία. Δεν επαναλαμβάνω την ψηφοφορία επειδή μου αρέσει το αποτέλεσμα. Απλά το επαναλαμβάνω γιατί δεν έλαβα υπόψη την ψήφο μια συναδέλφου που ήταν παρούσα. Δεν την υπολόγισα, δεν την μέτρησα. Λυπούμε, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με μια πληροφορία που έχω, αποφασίζει ο ε, πρόεδρος ε, αν ε, ε, επιτρέπεται κάποιος να ψηφίσει χωρίς κάρτα ψηφοφορίας ή είναι ο ε, βολευτής αυτός ο οποίος αποφασίζει. Εγώ νομίζω ότι ε, μόνο εσείς μπορείτε να αποφασίσετε αν ε, η κυρία Μπερές για παράδειγμα που δεν είχε την κάρτα μπορούσε να ψηφίσει και αφού το αποφασίσατε και η κυρία Ζόμερ το ίδιο έπρεπε να κάνει. Ευχαριστώ πολύ που με υποστηρίζετε λέει. Γιατί αφού πραγματικά έλαβα τις ψήφους της κυρίας Μπερές υπόψη έπρεπε να λάβω και της κυρία Ζόμερ. Ωραίο, θα το συζητήσουμε. Ο κύριος Λίζε έχω μια πήγουσα παράκληση προς την κυρία Περές. Κανονικά, στην Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος, ε, ε, όποιος δεν έχει κάρτα ψηφοφορίας δεν μετρά τη ψήφος του. Και η κυρία Πρόεδρος, παρόλα αυτά, σας επέτρεψε να αφήσετε, γι' αυτό δείξτε κάποια αυτοσυγκράτηση και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ψηφοφορία, κυρία Περές. Ναι, κυρία Πρόεδρε, εδώ υπάρχει κάποια σύγχυση, αλλά θα συμφωνήσω με την κυρία Μπερέ. Το θέμα δεν είναι να ξέρουμε, να δούμε αν μπορούμε να ψηφίσουμε με ή χωρί κάρτα. Ε, το θέμα είναι ότι η ψηφοφορία έκλεισε το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε και υπάρχει άρθρο του οικονομισμού που ορίζει ότι είτε έγινε λάθο είτε όχι, εφόσον έχει κλείσει το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία, δεν μπορεί κανεί να αναχωρεί. Εδώ λοιπόν κρυβόμαστε πίσω από το πρόβλημα τη ε, παρουσίαση όχι μια κάρτα. Το λέει το άρθρο 164 και το θέμα είναι να έκλεισε ή και ψηφοφορία. Ωραία. Άλλο κανεί, ο κύριο πίσω. Πρόεδρε, έχετε το δικαίωμα να αποφασίσετε εάν μια κάρτα ψηφοφορία θα καταμετράτε ή όχι ω ψήφο και έχετε αποφασίσει ότι η ψηφοφορία έκλεισε. Δεν γίνεται ο πρόεδρο να έρχεται και να λέει με πέντε μέλη του Κοινοβουλίου ε, αργότερα από την ψηφοφορία πέντε λεπτά ότι «Α, σας είδα» ή «Δεν σας είδα». Ε, άμα, δεν, σας ειδα αμα δεν κοίταζα προ τα κέντρα, δεν σα είδα καθόλου. Δεν θα σα είχα δει καθόλου. Δεν γίνεται μετά το κλείσιμο της ψηφοφορίας να πάτε πίσω. Ωραία. Κατάλαβα, κατάλαβα τι λέτε. Δεν ήρθε όμω η κυρία μετά την ψηφοφορία. Δεν την είχα δει. Δεν την είχα δει γιατί ύψωνε το χέρι τη. Το σήκωνε. Αλλά όταν ξαναψηφίσαμε δεν ήταν τόσο κοντά τα αποτελέσματα. Υπήρχαν πέντε ψήφοι διαφορά την πρώτη φορά. Οπότε εν τέλει δική σα είναι η ψηφοφορία. Εσείς ψηφίζετε καλή μου. Εσείς ξέρετε αν θα ψηφιστεί περί κατά. Τι θέλετε κύριε Μπερέ, να ε, κρυφτούμε πίσω από ένα λάθο που έγινε ότι δεν καταμετρήθηκε μια συνάδελφο και να αλλάξει το αποτέλεσμα. είστε τόσο αυστηροί με την προφορία. δεν ξέρω πόσε ψήφοι θα ήταν υπέρ. Λυπάμαι που ήταν τόσο κοντινά τα αποτελέσματα, αλλά υπήρχαν και άλλοι συνάδελφοι που ήθελαν να ψηφίσουν ε, και εγώ αποφάσισα να ψηφιστεί δεύτερη φορά. Δεν θα αλλάξω απόφαση. Να καταμετρώνται οι ψήφοι σωστά, κάντε όλη τη δουλειά σα. Είμαστε εδώ να ψηφίσουμε και όλοι έχουν δικαίωμα στην ψήφο. Δεν είχα δει την κυρία Ζόμερ και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Και είναι δικό σα το αποτέλεσμα. Εγώ δεν βγάζω δικά μου αποτελέσματα. Εσεί το βγάλετε τα αποτελέσματα ω βουλευτέ που ψηφίσετε σε αυτή την αίθουσα για κάτι. Μην κρύβεστε πίσω από ένα λάθος και προσπαθείτε να κερδίσετε μια ψηφοφορία που δεν είχε την πλειοψηφία εν τέλει. Λυπούμε πολύ. Θα ψηφίσουμε τώρα, εάν θέλετε. Εάν δεν θέλετε, εάν δεν θέλετε, ευχαρίστω. Τώρα όμως ψηφίζουμε για την συμβαστική F2. Κυρία Μπερές, σας παρακαλώ. Δεν ξέρω πώ θα κάνετε αυτά στην ε, Επιτροπή ΕΚΟΝ. Δεν είναι εδώ ο κύριο Γουαλτιέρη για να με καθοδηγήσει. Με συγχωρείτε, αλλά θα το κάνουμε όπω το κάνω εγώ. Εγώ προεδρεύω σε αυτή τη συνεδρίαση και δεν θα σα δώσω το λόγο ξανά. Λυπούμε. Λυπούμε. Τροπολογία F2. F2. Ψηφίζουμε για την F2. Ποιοι είναι υπέρ της F2. Κατά. Έλεγχος. And it's Πέρας. Η κυρία Μπερές δεν ψηφίζει, η κυρία Ζόμερ ψηφίζει εκείνη υπέρ. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβιβαστική FA. Υπέρ της FA. Κατά. Έλεγχος. And uh, it is, uh, so to be honest, I see για να είμαι ειλικρινής, βλέπω ότι πολλές κάρτες κυκλοφορούν, αλλά δεν ψηφίζετε όλοι. Σας το λέω. Εμένα θα μου τη φέρουν την κάρτα μου. No, no. I'm recovering my card. Just Εμένα θα μου τη φέρουν την κάρτα μου, δύο λεφτά. I'm recovering my card. Welcome. Hello. Nice for you to join us. Sorry. Yeah. Okay. How are you voting? Τι ψηφίζετε. Υπέρ. Πόσες ψήφους ανεφ κάρτας έχουμε, κυρία Ζόμερ, κατά. Οπότε αλληλεξουδετερώνεστε. Απορρίπτεται. FB. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. FB2. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. And it's closed and we have uh, vote against. Uh, ε, ψηφίζω κατά δύο υπέρ, ένας κατά. Δύο κατά μάλλον, ένας υπέρ. Ε, εγκρίνεται. Τροπολογία G. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. H. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άι, υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Άι. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας υπέρ, ένας κατά. Δύο υπέρ, ένας κατά. Χωρίς κάρτες. Πέρας. Απορρίπτεται. Άι, δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. J. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. K. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. K2. Υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. k 2 Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δύο υπέρ ένας κατά. Απορρίπτατα. Συμβιβαστική L. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Με συγχωρείτε. Επειδή απορρίφθηκε η ψηφοφορία, θα η τροπολογία θα πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά όλες τις τροπολογίες. 4.49, υπέρ. 4.94, συγγνώμη, υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4,95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4,96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4,97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4,98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική L υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. άριστη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. L2 υπέρ. Κατά. Έλεγχο για την L2. ψηφοφορία. Ένα υπέρ, δύο κατά λήξης εγκρίνεται. Συμβαστική μη. Μη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Δύο κατά ένας υπέρ λήξης. Απορρίπτεται. M2. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δύο υπέρ ένας κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική νη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30, σελίδα 30. Μη α. Υπέρ, κατά, έλεγχος. Άρχεται την ψηφοφορία. Ένας κατά, δύο υπέρ. Πέρας. Πενήντα έξι και πενήντα πέντε. Απορρίπτεται. NB. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. X. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Με συγχωρείτε. Όλοι ήταν κατά. 5.54 σε δύο τμήματα. Και το μεσαίο τμήμα. Περίεργο. Το πρώτο τμήμα καταπίπτει. Το δεύτερο τμήμα. Όχι, πρέπει να το ψηφίσουμε. Δεύτερο τμήμα της 554. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το μεσαίο τμήμα. στην 554. Καταπίπτει, τελικά καταπίπτει. Με συγχωρείτε πολύ. Πολύ θα μ' άρεσε να ψηφίζαμε ένα μεσαίο τμήμα. Θα ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου. 5.55. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Ω. Ω. Συμβαστική Ό. Ε, υπέρ, κατά, αποχές για να ελέγξουμε. Ένας κατά, ακτιψηφορία. Ε, Πόσοι υπέρ, Σα ήρθε η κάρτα σα. Ωραία. Ένα κατά, ένα υπέρ. Ε, λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Σελίδα 34. Πι. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κιού. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ένας υπέρ, ένας κατά. Πέρας, απορρίπτεται. Συμβαστική Q2 υπέρ. Κατά. Αποχές, έλεγχος για την Q2. Θα μπορούσα να κρίνω, αλλά δεν θέλω να έχω αμφισβητήσεις. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την R. Άρχεται η ψηφοφορία. Μία ψήφος υπέρ, μία κατά. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική. Α, πρέπει να ψηφίσουμε τις τροπολογίες που καλύπτονται αυτή. 123 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 646 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε τη λογική σκέψεις. Συμβαστική ΑΑ. Συμβαστική ΑΑ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Μία ψήφος υπέρ, μία ψήφος κατά, πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τις τροπολογίες που καλύπτονται από τη συμβαστική. 125 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική αβ2 υπέρ, κατά, Αποχές Απορρίπτωται. Συμβαστική. Α, πρέπει να ψηφίσουμε την 127 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτωται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτωται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 129. Πέρας. Μία ψήφος υπέρ, μία ψήφος εναντίον ίσως. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική αλφαβήτα υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μία ψήφο υπέρ, μία κατά, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 133 υπέρ, 33 λέει πρόεδρος, 134 διορθώνει, 134 υπέρ, κατά, Έλεγχος για την 134. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μία υπέρ, μία εναντίον. ΕΛΚ, έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ. Κάποιος παρακαλώ να βγάλει την κάρτα του. Είναι αφαιρέσουν την κυρία Ζόμερ τώρα, εντάξει. Ε, εγκρίνεται λοιπόν. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συγκεντρωθείτε και σηκώνετε τα χέρια σας. Η δεμή θα μετρά μόνο τα χέρια που βλέπω. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Έλεγχος για τη 2 άρχεται γιατί δύο. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται με την ίδια διαφορά. Συμβαστική AC υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασ... Τροπολογία 139 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική AD υπέρ. Κατά αποχές μάλλον εγκρίνεται αλλά ας γίνει ελέγχος. Είναι συμβαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Κυρία Ζόμερ, είσαστε κατά. Α, έχετε την κάρτα εν τω μεταξύ. Κυρία Μπερέζ, ψηφίζετε δυνατά στο χειρό. πάντα. Ωραία. Πέρασα. Και έχουμε και μία ψήφο υπέρ, άρα εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, AF ε, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 149 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 150 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 151, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Συμβαστική AG. Πέφτει, καταπίπτει. Συμβαστική AG υπέρ. Κατά. Ας γίνει ένας έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπομονή μαζί μου, δεν τα ξέρω τόσο καλά. Είναι περίπλοκος ο κατάλογος ψηφοφοριών. Πέρας και μία ψήφο της κυρίας Μπέρες υπέρ. Απορρίπτεται. Τοπολογίες. Τοπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τοπολογία 152 υπέρ. Α, καταπίπτει. Εντάξει, εντάξει. Συγγνώμη. Χρειάζομαι βοήθεια. Α, σε παρακαλώ. Λοιπόν, 154 υπέρ. Κατά. Ακούστε, ακούστε. Εδώ μας δεν πρέπει να ψηφίσουμε, η Βαλιέτ, έτσι λέει. Είναι συμβατή σαν προσθήκη. Πρέπει να ψηφίσουμε την 154. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 155 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 155 ψηφίζουμε πέρας μία ψήφος εναντίον. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική. Α Ήτα. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΙ υπέρ κατά έλεγχος για την ΑΙ. Και έχουμε και μία ψήφο υπέρ, πέρας, εγκρίνεται συμβαστική AJ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΚ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. AL ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την AL. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Και μια ψήφος υπέρ, πέρα ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΜΗ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική, ΑΝ υπέρ αποχές εγκρίνεται α όμικρον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε να ελέγξουμε ωραία ψηφίζουμε στις τροπολογίες 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Έλεγχος για την 179. 179. Πέρας. Μία ψήφος εναντίον απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 181 ή μάλλον 100 μαζί και οι δύο, 181-182 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος για την 184. Άρχεται η ψηφοφορία φιλελεύθεροι ήταν εναντίον. Κυρία Μπερές, μία ψήφος εναντίον. Πέρας, απορρίπτεται. Συμβαστική AP υπέρ. Κατά. Εγκρίνατε. Συμβαστική AQ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AR υπέρ κατά έλεγχος για την AR άρχεται. Κυρία Μπερές, υπέρ. Πέρας. Απορρίπτεται. 56-57 πάρουμε και την ψήφο της κυρίας Μπέρες υπόψη, 57-57 και απορρίπτεται. Τροπολογίες που καλύπτονται τώρα από τη συμβαστική AR. 18 τώρα, υπέρ. Κατά αποχές, έλεγχος για το 18. Άλλη μια ψήφο υπέρ έχουμε, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος για την 194 άρχεται μια ψήφος υπέρ πέρας απορρίπτεται 195 υπέρ παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας τόσο πολύ δεν σας βλέπω υπέρ κατά απορρίπτεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. σημαστική AS υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την AS άρχεται. Πέρας. Και μία ψήφος υπέρ απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη 19 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 198. Άρχεται. Πέρας. Δεν ψηφίζετε όλοι, το ξέρετε. Απορρίπτεται λοιπόν. 197 υπέρ. Κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αλλά ελέγξουμε την 197 ξεκινάει η ψηφοφορία βλέπω ότι έχετε στις εισδοχές της κάρτες σας αλλά δεν ψηφίζουν όλοι μια ψήφος επίσης υπέρ απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική αλφα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AV υπέρ κατά έλεγχος για την AV άρχεται. Και μία ψήφο υπέρ, πέρας, απορρίπτονται. Ψηφίσουν τις τροπολογίες 21 υπέρ, κατά. Έλεγχος για την 21 άρχεται. Και μία ψήφος υπέρ, πέρας. Απορρίπτεται και πάλι 207 υπέρ. 207 κατά. Αποχές απορρίπτεται 206 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 210 υπέρ κατά έλεγχος για τη 210 ξεκινάει Μία ψήφος εναντίον, πέρας, δεν ψηφίσατε όλοι, αυτή είναι η ζωή όμως, να κάνουμε, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, οι σοσιαλιστές δεν μου δείξαν τίποτα. Α, είσαστε υπέρ. Ας ελέγξουμε για την 22. Άρχεται. Πέρας. Και έχουμε και μία ψήφο υπέρ, εγκρίνεται. Συμβιβαστική AW, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ΑΧ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται α υπέρ κατά έλεγχος για την α ή άρχεται ψηφοφορία και μία ψήφος υπέρ πέρας εγκρίνεται ΑΖ υπέρ κατά αποχές. In favor, so it's adopted. Εγκρίνεται. 2.23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3α, α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα συμβαστική με 3β, β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα συμβαστική με τριπλό C υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε. Αυτό είναι για το Brexit. Ε. Λοιπόν, αυτό, αυτό τονίζει και ισχυροποιεί το Brexit. Συμβαστική με τριπλό D υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Για το τριπλό D. D, D, D. Άρχεται και μία ψήφος υπέρ, πέρας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τριπλό ε, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 242 υπέρ, κατά αποχές, έλεγχος για τη 242 άρχεται και μία ψήφος εναντίον. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τριπλό F υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος λοιπόν για το τριπλό F άρχεται. Η τελευταία σελίδα είναι παρακαλώ συγκεντρωθείτε. Τριπλό F. Ψηφίσατε όλοι. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε και μία ψήφος υπέρ. Δεν ψήφισαν όλοι. Ας κλείσουμε όμως. Με μία ψήφο υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 28. Άρχεται η ψηφοφορία και μία ψήφος υπέρ, πέρας, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζετε. Στην προηγούμενη δεν ψηφίσατε. Έξι από εσάς. Το σχέδιο της εκθέσεως ως ετροποποιήθη ηλεκτρονικά. Κύριε Eichhout, τι θέλετε να πείτε. Μπορούμε να έχουμε μισό λεπτό να ρίξουμε ματιά σε όλα τα αποτελέσματα. Ζητώ πέντε λεπτά για να δούνε όλες οι ομάδες τα αποτελέσματα. Κύριε Έκχαουτ, είστε εισηγητής, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τρία λεπτά να το κάνουμε, τρία. Πέντε, λέει και ο Σέικχαουτ. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να ικανοποιήσουμε το αίτημα ενός από τους εισηγητές. Παρακαλώ, κάνουμε μικρό διάλειμμα για κουβέντα, συζήτηση. Now for the final vote, if you are ready, people. Ο κύριος Κουαλτιέρη ήρθε στην παρέα μας. Επομένως, αυτός ε, θα κηρύξει την ψηφοφορία για την οριστική, την τελική ψηφοφορία. Να βάλετε το κερασάκι στην τούρτα, εσάς το άφησα, την τελική ψηφοφορία δεν ήταν και τόσο εύκολο να έρθω από, το, από τη Φραγκφούρτη, λέει ο κ. Γκουαλτιέρη. Τέλο πάντων, άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστικά ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορία. 52 ψήφοι υπέρ, 44 συν 1 κατά. 19 αποχές εγκρίνεται. So, thank you very, very much. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν όλες και όλους πέρα στη συνεδρίαση.